Μια ανακοίνωση τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι στη διαθέσή σα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνονται. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει λοιπόν. Και έχω λάβει από το Συμβούλιο.